Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έναρξη. Ξεκινάμε, ξεκινούμε την κοινή δημόσια κρόση για το θέμα του κράτους δικαίου. Θέλω να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων εκ μέρους της ΛΥΜΠΕ η ακρόαση για το κράτος δικαίου στη διαδικασία προς, ε, ε, θα μετα, μεταδίδεται διαδικτυακά και έχουμε το καθεστώς ε, της διερμηνίας που γνωρίζετε. Σήμερα θα επικεντρωθούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην πρόοδο και στι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιε χώρε για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κράτου δικαίου που σχετίζονται με τα ονομαζόμενα κριτήρια Κοπενχάγη. Όσον αφορά τον ε, σεβασμό των ε, αξιών του άρθρου 2 τη συνθήκη των συνθήκων υπάρχουν και υποχρεώσεις ε, των υποψηφίων χωρών με βάση τα κριτήρια τη Κοπενχάγης που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα κράτη-μέλη μετά την ένταξή του στην Ένωση. Η πρακτική έχει δείξει ότι η παρακολούθηση των κριτηρίων αυτών μετά την ένταξη μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Ω εκ τούτου, εδώ σήμερα θα μελετήσουμε πώ θα ενισχύσουμε τα θέματα και τη μελέτη των κεφαλαίων του κράτου δικαίου εν ώψη της ένταξης και πώ θα ενισχύσουμε τον πολιτισμό του κράτου δικαίου σύμφωνα με τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπω γνωρίζετε, θυμίσουμε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ήταν στο επίκεντρο πολλών δραστηριοτήτων και ε, πρωτοβουλειών σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Ένωση. Η αποκατάσταση σοβαρών ε, παραβιάσεων του κράτους δικαίου από κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη της διαδικασίας του άρθρου 7 που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια όλοι μας παρακολουθούμε όπως επίσης και το άρθρο 7 ε, προβλέπει και για κυρώσεις όταν γίνεται σοβαρή παραβίαση των αξιών. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη έχει υπάρξει στα θέματα της ημερήσιας δάταξης ε, και η κατάσταση του, σε σχέση με το άρθρο 7 που ξεκίνησε στην Πολωνία. Τον Ιούνιο του 2018 η Επιτροπή μας αποφάσισε να δημιουργήσει μια Επιτροπή Παρακολούθησης που θα έχει τη γενική εντολή να παρακολουθεί το θέμα της, ε, του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, συντάσσει εκθέσεις οι προτάσεις θα υποβληθούν στην επόμενη Ολομέλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλο και με μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με τις υπάρχουσες όσο πιθανές παραβιάσεις των αξιών, το Κοινοβούλιο ε, υιοθέτησε δύο, ψηφο, ψηφίσματα τον, ε, το 2016 και το 2018 που ζητά έναν αποτελεσματικό καθο, ε, μηχανισμό παρακολούθησης ε, του κράτους δικαίου και των θεμελιών δικαιωμάτων. Επίσης, περιμένουμε την ανακοίνωση για την περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου τις επόμενες ημέρες. Έτσι, χαίρομαι που έχουμε υψηλούς εκπροσώπους από τους, ε, από διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου το Συμβουλίο της Ευρώπης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Χαίρομαι που βρίσκεστε όλοι εδώ και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευθύς εξ αρχής σας είπα ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που από κοινού προεδρεύουμε και, ε, και ε, οργανώνουμε την ακρόαση αυτή με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και γι' αυτό το λόγο θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Thank you. Gracias. I will speak in Spanish. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά ο, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο Χαβιέρ Κούσο. Και από πλευράς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να καλωσορίσω όλους σε αυτή την κοινή ακρόαση μεταξύ Επιτροπής Λιμπέ και Επιτροπής ε, ΑΦΕΤ η συνεδρίασή μας ε, είναι πολύ επίκαιρη, διότι δύο εβδομάδες ε, μετά από την αποστολή δύο αντιπροσωπιών ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, η μία στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο και η άλλη στην Αλβανία και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πλέον Βόρεια Μακεδονία. Ε, οι περισσότερες είναι χώρες υποψήφιες, ε, πιθανή υποψήφια επίσης. Ε, η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι οι μόνες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης και η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία ελπίζουν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης φέτος. Η διαδικασία προσχώρησης περιλαμβάνει πρώτα τα βασικά και μετά στενή παρακολούθηση του κράτους ε, Εξακολουθούμε όμως να βλέπουμε κάποια αδράνεια και μια υπαναχώρηση θα έλεγα σε κάποια πράγματα, κυρίως ε, στις χώρες που είναι πρωτοπόροι, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο το κράτος δικαίου στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στην Τουρκία είναι πολύ ανησυχητικό και χαιρόμαστε που έχουμε προσκεκλημένους τόσο υψηλό επίπεδο εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να ρίξουμε και λίγο φως ε, στην όλη υπόθεση και να συζητήσουμε τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να αποφύγουμε αυτές τις επαναχωρήσεις. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να εκχωρήσω την Προεδρία στον κύριο Μωράης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κούτσο. Με τα χαρά σας σας παρουσιάσω την πρώτη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ξεκινάμε από τον κύριο Κρίστιαν Ντάνιλσεν που είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΑ. Επίσης έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζάνι Πουκιτσίο, πρόεδρο της Επιτροπής Βενετίας της Venice Commission του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ντάνιελσον. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Thank you. Uh, thank you. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συμπρόεδροι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ σήμερα να σας απευθύνω το λόγο για ένα θέμα το οποίο είναι σαφώς εντρεωμένος στις ε, σχέσεις μας με τις χώρες αυτές που είναι στον δρόμο της ε, διεύρυνσης. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, να εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό ε, πρώτα και μετά θα αναφερθώ στην προσέγγιση που έχουμε στην πράξη. Είναι σαφές ότι το κράτος δικαίου είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο γιατί σε αυτό βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται ξεκάθαρα στις ε, συνθήκες και αυτό ε, βεβαίως απαιτείται και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 49 της συνθήκης λέει ότι τα κράτη τα οποία ε, θέλουν να γίνουν μέλη της Ένωσης θα πρέπει να πληρούν αυτή τη συνθήκη, να προωθούν τις κοινέ αξίες και αυτές περιλαμβάνουν και το κράτος δικαίου. Και αυτό βεβαίως ε, υπάρχει και στα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης τα οποία απαιτούν ε, σταθερά θεσμικά όργανα, τα οποία σέβονται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Υπάρχει λοιπόν και μια πολιτική βούληση, η βούληση των πολιτών, αν θέλετε, στα Βαλκάνια, που θέλουν να ζουν σε χώρες οι οποίες θα ευημερούν και θα έχουν κράτος δικαίου και δεν θα υπάρχει διαφθορά και όπου θα είναι ανεξάρτητη και αποτελεσματική η δικαιοσύνη και η εξουσία θα αλλάζει μέσω εκλογών και ας είμαστε δικαίοι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και στις μεταρρυθμίσεις και στο να ξεπεραστεί η κληρονομιά του πολέμου και των συγκρούσεων στο Βαλκάνια αλλά ταυτόχρονα καμία από τις ε, χώρες περιοχής ε, δεν πληρεί τις ε, προϋποθέσεις για να γίνει μέλος και σε κάποιες δυστυχώς έχουμε δει μια στασιμότητα αν όχι και οπισθοχώρηση όπως είπατε κύριε Πρόεδρε οπότε απαιτούνται ακριβώς κάποια περαιτέρω στοιχεία για να υπάρξουν πιστικές μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική προσέγγιση της Κομισιόν. Από το 2012 έχουμε μία νέα προσέγγιση που βασίζεται στα μαθήματα που αντλούμε από τις μεταρρυθμίσεις αλλά και το ιστορικό της ε, κάθε χώρας και υπάρχει έτσι ένα ενισχυμένο σύστημα διαπραγματεύσεων με κάποια στη σημεία αξιολόγησης ε, με λεπτομερείς οδικούς χάρτες στα κεφάλαια 23 και 24, τα σχετικά κεφάλαια, ενδιάμεσους ε, στόχους και τελικούς στόχους. Υπάρχουν επίσης ε, κάποιες δικλείδες ασφαλείας, παραδείγματο χάρη στην περίπτωση καθυστερήσεων στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης και έτσι ώστε να υπάρχει μια γενικότερη ισορροπία η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να σταματήσει τις τεχνικές διαπραγματεύσεις σε άλλα κεφάλαια και στην χειρότερη περίπτωση όπως ε, σοβαρές και μόνιμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, ένα βασικό δίδαγμα από το παρελθόν είναι η σημασία του να κάνουμε πρώτα τα βασικά. Γι' αυτό το 2013 ε, ξεκινήσαμε αυτήν την προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι εστιάζουμε στα βασικά που περιλαμβάνουν το κράτος δικαίου, που σχετίζονται με τις βασικές αξίες και πλέον αυτή είναι ο κύριος πυλώνας ε, της πολιτικής μας ε, και η ενίσχυση και των δημοκρατικών θεσμών και η μεταρρύθμιση της δημοσίας και η ανταγωνιστικότητα βεβαίως και τα υπόλοιπα παραμένουν βασικές προτεραιότητες. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος δωρητής στην περιοχή, οπότε έχουμε έναν οικονομικό μοχλό πίεση ε, και το, το προενταξιακό μέσο του 2013 έχει έναν προπολογισμό 11,5 δισεκατομμύριων και το επόμενο μέσο που άρχισε να ισχύει το 2014 μέχρι το 2020 είχε 11,7 δισεκατομμύρια και προτείναμε για το τρίτο μέσο για την περίοδο 2021-2027 μια αύξηση 30% δηλαδή να φτάσουμε σε ένα ύψος 14,5 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε λοιπόν για σημαντικούς πόρους που έχουμε που ε, εστιάζουν και χρησιμοποιούνται κυρίως για αυτά τα βασικά. Από μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης μέχρι μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ε, μέχρι ζητήματα ενίσχυσης των κοινοβουλίων και των δημοκρατικών θεσμών για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Και Χρησιμοποιούμε και την ε, στήριξή μα ακριβώ ω εργαλείο για να τιμωρήσουμε την έλλειψη μεταρρυθμίσεων και να προωθήσουμε τη χρηματοδότηση τη κοινωνία των ε, πολιτών ε, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, την Τουρκία, όπου υπήρχε σημαντική μείωση των κοινοτικών επενδύσεων, ενώ μετατοπίστηκε η χρηματοδότηση σε αυτού που προωθούσαν τι αλλαγέ του κρατζοκαίου. Από το 2015 επίση, εφαρμόζουμε μια νέα μεθοδολογία για τις εκθέσεις πρόοδου για να ε, είναι πιο συγκρίσιμες οι αιτήσιε εκθέσεις. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε επιπλέον κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες θα είναι πιο ακριβείς. Και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια που θεωρούμε ότι είναι σημαντική από πολιτική σκοπιά για τις ε, Ενδιαφερόμενε χώρες. Δηλαδή είναι ευκολότερο να γίνει μια συζήτηση με βάση αυτές τις εκθέσει και θα διευκολύνει και την μεγαλύτερη εξέταση των μεταρρυθμίσεων από όλου του ενδιαφερόμενους στα κεφάλαια 23 και 24 και σε όλα τα κεφάλαια. Όπως είπα, δίνουμε σαφείς κατευθύνσεις για το τι αναμένουμε να είναι τα επόμενα βήματα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Και τέλος, τον Φεβρουάριο του 2018 η Κομισιόν δεσμεύτηκε για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων με την υιοθέτηση της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα ε, προσήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείξαμε ότι η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ανοιχτή, αλλά επίσης κατέστησε σαφές ότι δεν είναι μια επιταγή εν λευκό και απαιτεί μια λογική επιλογή από τους εταίρους μας, δηλαδή μια δύσκολη διαδικασία μετασχηματισμού και πράγματι αυτό σημαίνει διακυβέρνηση, κράτος δικαίου, αυτά τα οποία ανέφερα, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης και συμφιλίωση. Η διακήρυξη της Σόφιας επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα των καρτών μελών της Ένωσης για να εντείνουν τις επαφές σε όλα τα επίπεδα για να υπάρξει κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός μετασχηματισμός. Οπότε τα πρωτότυπα στοιχεία τα οποία προέκυψαν και αξίζει να τονίσουμε είναι ότι πηγαίνουμε πιο πολύ σε μια επιχειρησιακή συνεργασία στα θέματα κράτους δικαίου και αυτό σημαίνει παραδείγματο χάρη ένα πιο ισχυρό ρόλο για τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol, Eurojust κτλ. Επίσης περισσότερα εργαλεία παρακολούθησης ε, όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης με βάση και της Παγκόσμιας Τράπεζας και κάποιους δείκτες από το Συμβούλιο της Ευρώπης και στην καταπολέμηση της διαφθοράς επίσης μια παρόμοια προσέγγιση υπάρχει και στο οργανωμένο έγκλημα όπως το σχετικό έργο που έχουμε με τον ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των δικών. Και έχουμε επίσης αυξημένη στήριξη για την κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα ΜΜΕ να καταλήξουμε ένα παράδειγμα της ε, αυξημένης στήριξής μας για το κράτος και μετά από πολλές επενδύσεις για την νομική ευθυγράμμιση τώρα περνάμε προς πιο επιχειρησιακή βοήθεια και συνεργασία στο κράτος δικαίου και ήδη έχουμε αποτελέσματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Κομισιόν και την Γερμανία και το εκτελεί μια Ιταλο γερμανο-ολλανδική κοινοπραξία για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των δυνάμεων που παλεύουν στην πρώτη γραμμή το οργανωμένο έγκλημα και ως αποτέλεσμα είχαμε μία από τις μεγαλύτερες ε, συλλήψεις ε, ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια Μία 20 τόνους ε, χασίς που βρέθηκε σε ένα φορτηγό το οποίο κατασχέθηκε και συνελήφθη το πλήρωμα. Οπότε έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή, έχουμε αυστηρούς όρους, αλλά με δικαιοσύνη και εξετάζουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνει κάθε χώρα. Η εμπλοκή μας με την περιοχή αυτή είναι βεβαίως σήμερα πιο εντατική από ποτέ και με τα συμπεράσματα της Σόφιας ακριβώς τονίζουμε την σημασία αυτών των μεταρρυθμίσεων και τώρα επαφείται στι χώρε αυτές να έχουν κάποια αποτελέσματα και να δείξουν την αποφασιστικότητά τους και την πολιτική τους βούληση για μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στον Πρόεδρο της Επιτροπής της Βενετίας, τον κύριο Τζάνι Μπουκίκιο. Κύριε Μπουκίκιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε, Κυρίε και κύριοι. Η σημασία του κράτους δικαίου ως βασικό ορόσημο στη διαδικασία προσχώρησης είναι πλέον κάτι αδιαμφισβήτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου. Μόνο χώρες στις οποίες μπορούμε να περιμένουμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο θα εφαρμοστεί σωστά είναι κατάλληλες για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή της Βενετίας έχει ε, καταρτήσει έναν ε, έντυπο ελέγχου του κράτους δικαίου που καθορίζει κάποιες λεπτομέρειες για τα διάφορα στοιχεία του κράτους δικαίου. Αυτός το έντυπο ελέγχου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν εξετάζουμε την κατάσταση του κράτους δικαίου σε μια συγκεκριμένη χώρα και μπορούμε να κάνουμε μια διεξοδική, αντικειμενική, διάφανη και ε, ισότιμη αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτό το έντυπο ελέγχου, το checklist, μας δείχνει ότι το κράτος δικαίου δεν είναι ένα θέμα το οποίο περιορίζεται στο δικαστικό σύστημα. Απαιτεί επίση η διοίκηση, ε, η κυβέρνηση να δρά βάσει του δικαίου και όχι αυθαίρετα και ότι υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει για τη διαδικασία της νομοθέτησης. Αλλά στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα επικεντρωθώ στην ανεξαρτησία και στην αμεροληψία του δικαστικού ως το πιο βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου. Η ανεξαρτησία αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τα τακτικά δικαστήρια, αλλά και για τα συνταγματικά δικαστήρια. Τα συνταγματικά δικαστήρια έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την εγκαθίδρυση και την προάσπιση του κράτους δικαίου σε κάποιες υποψήφιες χώρες οι πολιτικοί συχνά μπαίνουν στον πειρασμό να επιτεθούν σε αυτά τα δικαστήρια όταν ε, εκδίδουν αποφάσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο ευπράσδεκτες σε όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας. Εγώ προσωπικά επανελειμμένος χρειάστηκε να προσπίσω το, το γεωργιανό, το τουρκικό και άλλα συνταγματικά δικαστήρια ε, και εκτός Ευρώπης ε, κατά επιθέσεων από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της χώρας. Ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε όλο ένα και περισσότερο μια λαϊκιστική τάση η οποία ισχυρίζεται ότι το να κερδίσει κανείς τις εκλογές δίνει το δικαίωμα στην πλειοψηφία να κυβερνά χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτή η νοοτροπία του ο νικητής τα παίρνει όλα είναι επικίνδυνη για το κράτος δικαίου. Τα σταυματικά δικαστήρια είναι τα όργανα τα οποία πρέπει να ε, προσδίδουν μια ισορροπία μεταξύ του κανόνα της πλειοψηφίας και της προστασία της μειοψηφία. Και πρέπει να τα βλέπουμε ω τέτοια και να τα υποστηρίζουμε σε αυτό το ρόλο. Όσον αφορά τα τακτικά δικαστήρια, το Συμβούλιο τη Ευρώπη, όπω επίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πτώση του τείχου του Βερολίνου και μετά έχουν κάνει τεράστιε προσπάθειε για να ενισχύσουν το δικαστικό στι χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώ και στην Τουρκία. Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι σε αρκετέ χώρε τα αποτελέσματα που επετέφθησαν ήταν απογοητευτικά. Το δικαστικό σύστημα αποδείχθηκε ότι είναι ένα τομέα πολύ δύσκολο να μεταρρυθμιστεί. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι 30 χρόνια μετά το τέλος του κομμουνισμού ε, η κατάσταση του δικαστικού συστήματος ε, σε μετακομμουνιστικές χώρες εξακολουθεί ε, να μην επαρκεί. Και θα πρέπει καταρχάς να αναγνωρίσουμε ότι αυτό κυρίως δεν οφείλεται σε κακούς κανόνες ή σε έλλειψη νομικών κανόνων. Όλες οι νέες δημοκρατίες έχουν ε, ε, προσυπογράψει τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας ε, στο Σύνταγμά τους. Υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο και εμεί στην Επιτροπή της Βενετίας κάνουμε πολύ σκληρή προσπάθεια για την βελτίωση. Αλλά σε γενικές γραμμές οι κανόνες δεν είναι χειρότεροι από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Το πραγματικό πρόβλημα δεν έγκυται κυρίως στους νομικούς κανόνες. Η νομική νοοτροπία της χώρας και η νοοτροπία των νομικών ε, είναι πολύ πιο σημαντική από τους επίσημους κανόνες. Όταν ξεκίνησαν οι μεταρρυθμίσεις στη δεκαετία του 90, κατά πάσα πιθανότητα υποτιμήσαμε τη σημασία της νοοτροπίας ή πιστέψαμε ότι οι νεότερες γενιές ε, νομικών αυτομάτως θα ανέπτυσαν μια ε, νοοτροπία η οποία θα ήταν ευθυγραμμισμένη με το κράτος δικαίου. Επίσης, μπορεί να υποτιμήσαμε και τους δισταγμούς των πολιτικών να δεχθούν ότι τα ανεξάρτητα δικαστήρια μπορεί να λάβουν αποφάσεις αντίθετες στις επιθυμίες τους. Επιπλέον, το δικαστικό είναι τμήμα ενός δημοκρατικού κράτους. Ε, είναι υπόλογο στην κοινωνία. Και αυτό αυτή η λογοδοσία θα πρέπει να αντανακλάται και στη σύνθεση των ε, συμβουλίων που πρέπει να περιλαμβάνουν και ένα ισχυρό δικαστικό στοιχείο, αλλά και ε, απλούς πολίτες, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ένα τέτοιο σώμα δεν θα είναι απλώς ένα όχημα για να εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα. Κατά την ε, κατάρτιση και αξιολόγηση κανόνων χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα εστιάζει στην ανεξαρτησία αλλά δεν θα παραμελεί και τη λογοδοσία. Η φοιτεία των δικαστών μέχρι την ηλικία συνταξιοδότηση είναι κατά πάσα πιθανότητα και η πιο σημαντική εγγύηση τη δικαστική ανεξαρτησία. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να πρέπει να δεχτούμε κάποιε εξαιρέσει σε κάποιου βασικού κανόνε, όπω συνέβη στην Αλβανία. Μετά από την ε, παρουσίασή μου θα ακολουθήσει μια παρέμβαση για την Αλβανία όπου υπάρχει ευρύτατη διαφθορά και αυτό συνέβη ότι χρειάστηκε να υπάρχει ε, ένας γενικότερος έλεγχος των δικαστών εν ενεργεία. Η Επιτροπή της Βενετίας δέχτηκε αυτή την ανάγκη, ε, υπόκειται βέβαια σε συγκεκριμένε εγγυήσεις και χωρίς την θετική μας αξιολόγηση τα αλβανικά δικαστήρια κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαν προχωρήσει με τη διαδικασία και θα την είχαν πατάξει πρέπει να έχουμε μια πολύ προηγμένη προσέγγιση που θα έχει μια ισορροπία μεταξύ ανεξαρτησίας και λογοδοσίας και ισορροπίας μεταξύ σεβασμού των διεθνών προτύπων και την ανάγκη να προσαρμόσουμε τους κανόνες ανάλογα με την κατάσταση στην κάθε χώρα. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται οι κανόνες, θα πρέπει να συνεχίσουμε και να ε, ε, επιταχύνουμε την στήριξη που παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνατότητες του δικαστικού στις υποψήφιες χώρες για να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει διεθνών προδιαγραφών. Τέλος, δεν θα πρέπει να ε, ξεχάσω να αναφέρω και τους άλλους παράγοντες στο δικαστικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, εισαγγελείς και νομικούς. Οι εισαγγελείς μπορεί να είναι όργανο καταπίεσης της κυβέρνησης, αλλά μπορεί να είναι και οι μόνοι παράγοντες που θα είναι σε θέση να δράσουν κατά χρήσεων από αυτούς που κατέχουν την εξουσία και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στις πολιτικές τάξεις οι νομικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν ε, υποθέσεις στα δικαστήρια που ίσως δεν είναι τόσο επιθυμητές και να υπερασπίζονται αποτελεσματικά αυτούς οι οποίοι ε, διώκονται αδίκως. Πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ε, το να υπερασπίζονται ανθρώπους που θεωρούνται εχθροί του κράτους δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και αυτοί εχθροί του κράτους όπως συμβαίνει στην Τουρκία. Για να συνοψίσω, η κατάσταση του κράτους δικαίου θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στην απόφαση του κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή μια χώρα ως ε, κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτό, ωστόσο, ποτέ δεν θα είναι εύκολη απόφαση, διότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ε, σπανίως είναι άσπρο ή μαύρο. Αφενός, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μόχλευση που τη παρέχεται από τη διαδικασία προσχώρηση για να πιέσει τι υποψήφιε χώρε να προωθήσουν όσο περισσότερο το κράτο δικαίου όσο ε, γίνεται και από την άλλη η προοπτική της ε, ε, προσχώρησης πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη για να μην αποθαρρύνει χώρε από τι περαιτέρω προσπάθειε. Αυτό που θα θέλαμε να κάνουν οι κυβερνήσεις ε, σε υποψήφιες χώρες και να κατανοήσουν είναι ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα όχι για να ικανοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουν αποδεκτά ως μέλη, αλλά ε, ε, προς όφελος των πολιτών τους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε στην Αλβανία και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Έχω τη χαρά να δώσω το λόγο στον Τέο Γιάκοψ, ο οποίος είναι παρατηρητής ε, της Διεθνούς Επιχείρησης ε, Παρακολούθησης ε, της IMO στην Αλβανία που συνδράμει τις αρχές στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και υποστηρίζει τη διαδικασία της προσωρινής αξιολόγησης δικαστών και εισαγγελέων στην Αλβανία. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά το πολύ κύριε Γιάκοψ. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ καταρχήν για την ε, πρόσκληση στους διεθνείς παρατηρητές να παρευρεθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μοιραστούν μαζί σας αυτά που καθημερινά αντιμετωπίσουμε. Οι διεθνείς παρατηρητές στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης ε, παρακολούθησης είναι σε θέση να μεταφέρουν μια ε, σημαντική ε, και άνευ προηγουμένου άσκηση, επιχείρηση που πραγματοποιείται στην ε, Αλβανία έτσι ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί σωστά, σωστά το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και εκπροσωπώ και τους συναδέλφους μου. Έχω προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες, χωρί όμω πάρα πολλέ πληροφορίες. Πρώτη διαφάνεια. Ποια είναι η κατάσταση πριν από τον ε, έλεγχο αυτό στο δικαστικό χώρο της Αλβανίας. Ε, οτιδήποτε και αν ρωτήσετε θα βρείτε τρία βασικά στοιχεία. Εκτεταμένη διαφθορά, έλλειψη ανεξαρτησίας, πολιτική επιρροή και επίσης σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τις εγκληματικές ομάδες. Ε, μπορείτε να προσθέσετε και ένα τέταρτο στοιχείο που είναι μία συζητήσιμες ε, νομικές δεξιότητες και ικανότητες τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν προ του ελέγχου. Είναι απολύτω λοιπόν σαφές ότι οι πολίτες της Αλβανίας αντιμετώπισαν ένα ελληματικό δικαστικό σύστημα ε, και σαφώς το κράτος δικαίου δεν μπορούσε ούτε να λειτουργήσει σωστά ούτε να κάνει αυτά που έπρεπε. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο πάντα της ενόψη της, της πορείας προς την ένταξη αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια, ένα σύστημα επανεξέτασης των δικαστών, των εισαγγελέων και κάποιων τουλάχιστον ε, των, ε, από τους νομικούς συμβούλους στην Αλβανία τα, οι στόχοι και οι, τα αίτια αναφέρονται στο, σε ένα ε, άρθρο του ε, συντάγματος. Η επανεξέταση του συστήματος θα λειτουργήσει με σκοπό την την... Ε, να υπάρξει εγγύηση για τη σωστή λειτουργία του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, όπως επίσης και την επαναδημιουργία, την επαν... επανεγκατάσταση της ε, εμπιστοσύνης, της κοινή γνώμης προς αυτούς τους θεσμούς. Αυτά με δύο λόγια. Ε, έχω Σας έχω παρουσιάσει τα προβλήματα ή τα ελλείμματα που μπορούν να βρεθούν, μπορεί να βρει κανείς στο δικαστικό σύστημα της Αλβανίας. Δεν μας εκπλήσει ότι το πεδίο αυτού του ελέγχου στηρίζεται σε τρία βασικά κριτήρια, δηλαδή μια αξιολόγηση των, της υφιστάμενης κατάστασης, μια αξιολόγηση της προέλευσης και μια αξιολόγηση ικανότητας. Ε, αυτό μπορεί να γίνει σωστά μέχρι το ερώτημα τα στοιχεία των ε, δικαστών, των ε, εισαγγελέων και των νομικών συμβούλων συνάδουν με τα οικονομικά μέσα που μπορούν να δικαιολογήσουν και να εξηγήσουν ε, με, με εύλογα οι άνθρωποι αυτοί. Ο έλεγχος προέλευσης είναι εάν υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα σε αυτό το προσωπικό και, τις, ε, και παράνομες ομάδες ή ανθρώπους που εμπλέκονται στο ε, οργανωμένο έγκλημα και η ικανότητα ε, αξιολόγησης ε, ικανότητας έχουν πράγματι τα προσόντα να λειτουργήσουν ως δικαστές, εισαγγελείς και νομικοί σύμβουλοι. Αυτό έχει γίνει σε οκτώ περιπτώσεις, τρεις από τις οποίες προβάλλει ο κάθε ελεγχόμενο μόνος του και άλλες οι οποίες προκύπτουν από έρευνα ή διακλήρου. Ποιος κάνει το έργο αυτό. Τρεις οργανισμοί ελέγχου υπάρχουν κυρίως πρώτον η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Προσόντων, Ανεξάρτητη Επιτροπή Καταλληλότητας, που αποτελείται από τέσσερα σώματα τριών ε, επιτρόπων με, που αλλάζουν με πενταετή θητεία που θα λήξει το 2022. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το όργανο αυτό είναι ερευνητικό όργανο και στο τέλος της έρευνας τα αποτελέσματα αναφέρονται στους δικαστές εισαγγελείς και νομικούς, δηλαδή πρέπει και κατόπιν πρέπει αυτοί να φέρουν το βάρος της απόδειξης. Δηλαδή αν υπάρχουν αμφιβολίες τότε οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να φέρουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις κατηγορίες και η Επιτροπή ε, αποφασίζει σχετικά με την επιβεβαίωση ή την παραπομπή ή την ε, ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση. Το δεύτερο σώμα που συμμετέχει εδώ είναι οι δύο δημόσιοι επιτροποί εκπροσωπούν το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον και μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσόντων μετά από σύσταση των διεθνών παρατηρητών ή μπορούν και να το κάνουν και ε, εξοφίτσιο. Απλώς θέλω να σας πω ότι τα μέλη των διαφόρων αυτών οργάνων ελέγχου έχουν επιλογή και εκλεγή από το Κοινοβούλιο. Το τρίτο όργανο ελέγχου είναι ένα ειδικό εργαστήριο, ε, δικαστήριο ε, το οποίο είναι εφετείο, αποτελείται από επτά δικαστές με 9 ετή θητεία, είναι μέρος του, ε, είναι μέρος του συνταγματικού δικαστηρίου και οι ε, θέσεις αυτές, οι προσφυγές αυτές γίνονται μετά από ε, συνομιλίες και υποδείξεις ε, των διαφόρων οργάνων. Τώρα, η διεθνής εποπτεία. Η διεθνής κοινότητα έχει ξεκινήσει την ε, λεγόμενη επιχείρηση, ε, διεθνή επιχείρηση παρακολούθησης, όπου υπάρχουν οκτώ διεθνείς παρατηρητές, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, όπου εργαζόμαστε με 60 περίπου μέλη προσωπικού. Στόχος είναι η υποστήριξη και επανεκτίμηση της διαδικασίας με την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαδικασίας. Δεν καθοδηγούμε, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε να, καθοδηγήσουν, να καθοδηγηθεί λίγο η διαδικασία έρευνας. Στο διάστημα αυτής της ε, διερευνητικής φάσης μπορούμε να υποβάλουμε προσφυγές, συστάσεις, απόψεις εάν θεωρήσουμε ότι οι αποφάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής δεν είναι ε, απόλυτα σωστοί και μπορούμε να συμμετέχουμε αυτόν τον τρόπο. Συμμετέχουμε και στις συζητήσεις, δεν συζητούμε εμείς, αλλά παριστάμεθα και αφού ληφθεί η απόφαση μπορούμε να διατυπώσουμε τις διαφωνίες μας. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν οι διεθνείς παρατηρητές δεν ε, καθόμαστε εκεί απλώς για να παρακολουθήσουμε. Ε, έχουμε ενεργό ρόλο, συμμετέχουμε, εμπλεκόμεθα ε, ενεργά στην όλη αυτή διαδικασία ελέγχου. Για τον λόγο αυτό έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να κάνουμε αυτό που πρέπει, να διεκπαιρεώσουμε το ρόλο μας και πρέπει να σας πω ότι ε, η διαδικασία ελέγχου ε, δεν είναι απλώς επιφανειακή. Υπησέρχεται, προχωρεί σε βάθος και ασχολά, και α, τίθεται και το θέμα της ε, ιδιωτικότητας Τώρα όσον αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου μέχρι τώρα και για να υπογραμμίσουμε ότι η όλη αυτή διαδικασία πραχωρεί σε βάθος, πρέπει να πω ότι στον πρώτο βαθμό μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 111 υποθέσεις, 18 σε, επίπεδο, ε, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και 48 άτομα επιβεβαιώθηκαν και παραμένουν που σημαίνει ότι οι μισή περίπου έχουν ε, απολυθεί που είναι μεγάλο ποσοστό. Έχουμε 17 παρετήσεις. Ε, πρέπει να πούμε ότι αυτά συνάδουν με τις ε, απολύσεις γιατί οι πολλές από τις παρετήσεις είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να πούμε ότι το συνταγματικό δικαστήριο θα έπρεπε να αποτελείται από εννέα δικαστές ε, μόνον ένας δικαστής επιβεβαιώθηκε, παρέμεινε στη θέση του, οκτώ απολύθηκαν. Το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει να αποτελείται από 18 δικαστές, μόνο τρεις από αυτούς ε, παρέμειναν στη θέση τους, ε, οι υπόλοιποι ε, απομακρύνθηκαν. Και αυτό για να σας δείξω πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, τι μάθαμε, ε, ποια είναι η εμπειρία μας από αυτές τις πρακτικές. Αν θέλει κανείς να προχωρήσει εντελεχώς, συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο. Η δικαστική εξουσία είναι από τους πυλώνες του δημοκρατικού κράτους. Δεν το κάνει κανείς αυτό με κάποιες δευτερεύοντες νόμους. Χρειάζεται το θέμα αυτό να είναι ενσωματωμένο ενσωματωμένο στο ε, στο Σύνταγμα και να υπάρχουν και οι απαραίτητες εξουσίες αλλά και τα μέσα, τα εργαλεία για την εκτέλεση των εξουσιών αυτών. Τα εθνικά, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθοδηγούν αλλά χρειάζεται ε, έντονη διεθνής παρακολούθηση γιατί ε, χρειάζεται ε, και για την νομιμοποίηση όλων αυτών να ε, οι εργασίες να πραγματοποιούνται από, σε εθνικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται η εποπτεία και ο έλεγχος και βάση περιπτώσει να προσφέρεται υποστήριξη και συμβουλές και να προσπίζονται, να υπάρχει πρόσπιση των εθνικών φορέων. Τέλος, η διαδικασία αυτού ελέγχου που γίνεται με αυτόν τον τρόπο χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται επίσης πολύ ξεκάθαρη, σαφή προετοιμασία όχι μόνο επιχειρησιακά, δηλαδή ε, χώρος ε, ή προσωπικό αλλά και κριτήρια και διαδικασίες. Στο σενάριο αυτό δεν υπήρχε τίποτα που θα δεν προϋπήρχε κάτι που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Χρειάστηκε να κάνουμε μεγάλη προετοιμασία και αυτό ε, το συνιστούμε και στο μέλλον. Μακρά προετοιμασία είναι απολύτω απαραίτητη. Αυτό που είναι επίση πολύ χρήσιμο είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, ούτω ώστε να ε, ενημερωθούν οι πολίτες, η κοινή γνώμη για το τι είναι αυτός ο έλεγχος, χρειάζεται να εξηγηθεί όλη η διαδικασία και κυρίως να ε, γίνει σαφέ το τι δεν είναι, περί δεν πρόκειται αυτή η διαδικασία. Επίσης, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό το οποίο μάθαμε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν επιτόπου οι ρυθμίσεις για διεθνή νομική συνεργασία. Αυτή η διαδικασία ελέγχου δεν είναι ποινική διαδικασία. Έχουμε πολλά μέσα, αλλά πρέπει να έχουν γίνει απαραίτητες ρυθμίσεις. Επίσης, μέτρα αποκατάστασης πριν ξεκινήσει αυτή καθε αυτή η διαδικασία ελέγχου. Ε, λυπάμαι που ε, ξεπέρασα το χρόνο μου. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά μαθήματα, η μεγαλύτερη εμπειρία και οι βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώσαμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον ομιλητή. Προχωρούμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, ακρόασης αυτής, δηλαδή τον ε, μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του κράτους δικαίου και ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Μάρκο Κάμιτς που είναι εκπροσωπεί το Κέντρο Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου του Γράτ στην Αυστρία. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά το πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπρόεδροι, από τα μέλη της Επιτροπής, ε, κυρίες και κύριοι, ήδη ακούσαμε πως η αιρεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου συνεχώς αναβαθμίζεται και έχει πολλές δυνατότητες για την μεταρρύθμιση των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Παρ' όλα αυτά, ο αντίκτυπος της ε, παραμένει περιορισμένος και φαίνεται πως αντί να ενισχύει τις ε, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις φαίνεται ότι η δημοκρατία υπαναχωρεί στα Δυτικά Βαλκάνια ενώ ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων είναι αργός και οι ε, μεταρρυθμίσεις ακόμα δεν ε, έχουν εδρεωθεί και περιέργως αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενταξιακή διαδικασία. Οπότε τι μαθήματα βγαίνουν από αυτό και τι συστάσεις ε, μπορούμε να κάνουμε. Θα εστιάσω σε τριών ειδών συστάσεις. Ε, πρώτον, την ανάγκη βελτίωσης των εργαλείων της, εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση και τις εκθέσεις δεύτερον για την ρύθμιση της οικονομικής στήριξης των χωρών της περιοχής έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα κίνητρα και οι κυρώσεις ε, και τέλος η ανάγκη να γίνουν αυτά τα ζητήματα όχι απλώς ε, μια διαδικασία νομική ή τεχνοκρατική αλλά μια κοινωνική η οποία θα προκύπτει από τις ίδιες τις ε, κοινωνίες και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι δυνατότητε των διαπραγματεύσεων δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα θέλαμε γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη κατεύθυνση θα έλεγα προς τον στόχο της ένταξης οπότε έτσι δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίε των ελλείψεων του κράτους δικαίου δηλαδή αυταρχικός τρόπος διακυβέρνησης έχουμε ισχυρούς άντρες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για μεταρρυθμίσεις αλλά θέλουν να διατηρήσουν το status quo, αλλά και τα, μηνύματα με που έρχονται από τις Βρυξέλλες είναι ασαφή και ενθαρρύνουν του ε, τους ε, κρατούντες. Ε, δεύτερον, κάποιοι πιθανώς ισχυροί μηχανισμοί που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορές ρήτρες παραδείγματος χάνει, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου και να έχετε κατανοητή ότι το Μαυροβούνιο απέχει μόνο ένα κεφάλαιο ακόμα να ολοκληρώσει οπότε δεν ξέρουμε τι ε, επιτυχία θα έχει ο μηχανισμός αυτό στο μέλλον και τέλος υπάρχει η έννοια αυτή της ε, σταθερότητας ε, που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αγνοεί την υπαναχώρηση της δημοκρατίας οπότε τι ακριβώς μπορεί να γίνει όταν μιλάμε για αυτές τις αποστολές ε, επανεξέταση και παρακολούθησης. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά τα ζητήματα μένουν ε, στα χαρτιά και τα είπε και ο συνάδελφός μου, η κυρία Μάρκ, και αυτό φαίνεται από το ότι η διαδικασία αυτή υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, αλλά ακόμα και οι ειδικοί ελάχιστα γνωρίζουν με την εξαίρεση της έκθεσης Πρίμπε του 2015 τι έχει λοιπόν το ιδιαίτερο η έκθεση Πρίβε που ασχολήθηκε με την Βόρεια Μακεδονία. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια συγκεκριμένη έντολη για να αναλύσει γρήγορα ζητήματα που προέκυψαν από κάποια σκάνδαλα υποκλοπών που έγιναν στην ε, χώρα και βέβαια υπήρχε μια πολύ τεταμένη κατάσταση που επίσης σχετίζεται με τα όσα βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, υπήρχε άμεση σχέση του πλαισίου της αποστολής ε, και της επιδίνωσης του κράτους δικαίου. Τέταρτον, είχε μια εντολή να κάνει συστάσεις για συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση της χώρας ε, και τέλος ε, υπήρχε πλήρης στήριξη από μια ομάδα ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την αποστολή στη χώρα. Επίσης, θα ήθελα να πω πως η έκθεση Πρίμπε τότε αποκάλυψε ότι φαίνεται ότι δεν υπήρχε επαρκή γνώση για τα ζητήματα που αποτελούν το αντικείμενο της αποστολής. Ποια είναι τα συμπεράσματα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα η εντολή για επανεξέταση από μοτιμούς θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη χρονικά με συγκεκριμένες ε, διορίες. Δεύτερον, δεδομένης ε, της ε, πολύ μικρής προθεσμίας, καθώς θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε τρεις μέρες επιτόπου, θα πρέπει να υπάρχει μια εκτενή προετοιμασία. Και τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία έτσι ώστε οι οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να παρακολουθούν την ε, πρόοδο και βεβαίως ε, και η δημοσιοποίηση των ονομάτων των συντακτών των εκθέσεων θα σημαίνει και μεγαλύτερη αξιοπιστία όπως έγινε και με την έκθεση πριν. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις εκθέσεις σημασία έχει να μην σιωπούμε η φωνή της Κομισιόν πρέπει να ακουστεί περισσότερο γιατί αν δεν μιλάει για τις παραβιάσεις ανθρωπίνου δικαίου και της, ε, την διάβρωση της δημοκρατίας ή εκστρατείας λάσπης ε, κατά των ΜΜΕ και των λοιπόν ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους διαφορούς αυταρχικούς κυβερνώντες να συνεχίσουν να κάνουν τα όσα κάνουν και πάλι δεν υπάρχει κάποια συνέχεια που να δίνεται σε αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε σε ε, non-paper για τέτοια ζητήματα. Οπότε, όταν μιλάμε επίση για την συγκριτική αξιολόγηση, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται πέρα από την ε, τεχνοκρατική ε, φάση και θα πρέπει να εστιάζει ακριβώς σε αυτές τις ελλείψεις της δημοκρατίας. δηλαδή να εκθέτει την πρόοδο ή την ε, έλλειψη προόδου μέσω ενός υποδείγματος ε, για να υπάρχει και ένας ε, φιλικός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων χωρών και μια ετήσια ανασκόπηση της προόδου και κάποια κίνητρα αλλά και κυρώσεις. Δεύτερον, Και εδώ πέρα οφείλω να συγχαρώ την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και όλους τους ε, εμπλεκόμενους ε, στο προενταξιακό μέσο 3 που προβλέπει την διακοπή σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης ε, του κράτους δικαίου. Αλλά πρέπει επίσης να δούμε και κάποιες από τις δυσλειτουργίες του δεύτερου προενταξιακού μέσου ότι δηλαδή θεωρούν ως υπόδειγμα τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια κάτι το οποίο είναι θετικό, αλλά υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να υπάρχει αυτή η στήριξη να μην υπάρχει στήριξη, με συγχωρείτε, για έργα τα οποία δεν στηρίζονται από το κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή την οικονομική στήριξη της Κομισιόν. Και τέλος, όταν μιλάμε για την ανάγκη αύξηση ε, της πίεση όχι μόνο από πάνω γιατί μέχρι στιγμής γι' αυτό μίλησα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους ε, πολιτικούς των Βαλκανίων αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος ε, που επίσης θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη στήριξη μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων και της εμπειρίας της κοινωνίας των πολιτών από κοινού με τις κυβερνήσεις των Δικών Βαλκανίων που θα πρέπει να είναι η βασική σύμμαχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε η πολιτική ηγεσία ε, των χωρών της περιοχής να έρθει πιο κοντά στις ε, προδιαγραφέ του κράτους δικαίου και να μπορέσουν έτσι οι χώρες να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια κοινωνική αλλαγή όπως είπα στην αρχή δηλαδή θα χρειαστεί γενιές γιατί αν εστιάσουμε μόνο στην αλλαγή των νόμων και των θεσμικών οργάνων ε, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα οπότε αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία, να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ε, να ελέγχονται οι, οι πολιτικές ηγεσίε για να έχουν κίνητρο να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και όχι να διατηρήσουν το status quo και μόνο μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητα για να είναι υπόλογες οι ελίτ ε, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ένταξης αλλά και μετά την ένταξη καθώς έτσι την διαδικασία αυτή μη αναστρέψιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα έχουμε τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Ρασίντ, εκτελεστικός διευθυντής ε, του ερευνητική ομάδας για τα Βαλκάνια στην Πριστίνα. Αγαπητοί Πρόεδροι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω όλες τις πλευρές και τις δυσκολίες που οδηγούν ε, στο κράτος δικαίου ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά θα ήθελα και να μεταφέρω την πλευρά της κοινή γνώμης του κόσμου. Τι σκέφτεται ο κόσμος. Πρώτον, η ε, ένταξη και η ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασική όρη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου πάρα πολύ απίθανο θα ήταν να πραγματοποιηθούν στα Δυτικά Βαλκάνια εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου εν ώψη της προπτικής της ένταξης. Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μάθει ε, ποιο είναι ο στενός δεσμός των ε, εσωτερικών και των περιφερειακών θεματολογίων με την ευρωπαϊκή ένταξη και νομίζω και οι πολίτες θα, το έχουν, το, ε, θα ε, έχουν συνειδητοποιήσει το ίδιο πράγμα. Θα το, θα το σαφώς δοκιμάσει σύντομα και η Μακεδονία. Δεύτερον, υπάρχει και ένα αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια, στην κατανόηση και την έκφραση του νοήματος των μεταρρυθμίσεων. Πριν από μερικά χρόνια και οι δύο είχαν μια πιο ε, συγγενή άποψη σχετικά με το τι θα σημάνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα οι διαφορές είναι πολύ ευρύτερες. Υπάρχει ένα ξανόμενο χάσμα για το, από τον τρόπο με τον οποίο ε, ερμηνεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια ε, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, το νόημά τους, πώς τις αξιολογούν, πώς τις εφαρμόζουν και ποιε είναι οι επιπτώσεις τους. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό κατά την άποψή μου και ισχύει κυρίως τώρα ε, στην περίπτωση της Σερβίας, του Κωσυφοπεδίου και της Αλβανίας. Σε κάποιες περιπτώσεις η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στα χαρτιά επιδεινώνει μόνο την κατάσταση. Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μάθει πώς να ξεγελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειλικρινά μερικές φορές τα στελέχη της Ένωσης γνωρίζουν ότι τους ξεγελούν και έχουν κάποιες δυσκολίες στην πολιτική ατζέντα τους ώστε ε, πολύ συχνά να διαφοροποιούν τις προτεραιότητές τους. Βεβαίω αυτή είναι η πραγματικότητα των Δυστικών Βαλκανίων ε, και η επίλυση των πολιτικών ε, ε, διαφορών και των λεπτών συγκρούσεων και διαφωνιών και επίσης η μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσουν εκ παραλλήλου. Ο ρυθμός της προόδου και στους δύο τομείς θα έπρεπε να είναι ταχύτερος από ό,τι διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια. Και επίσης σε γενικές γραμμές υπάρχουν βασικοί ηγέτες που δεν μπορούν μπόρεσαν να, ε, έχουν, να είναι αποτελεσματικοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ε, πολίτες τους. Η, Βόρεια Μακεδονία έδειξε ότι μπορεί να κάνει και τα δύο τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η καλύτερη περίπτωση, ο καλύτερος μαθητής ε, από, τα, όλα, όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα υπάρξει καλύτερο ε, καλύτερη περίπτωση. Η Σερβία δεν θέλει να τα κάνει και τα δύο. Η ηγεσία χρησιμοποιεί ε, τα πολιτικά θέματα για να υπονομεύσει τις προσπάθειες ε, μεταρρύθμισης και του κράτους δικαίου και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει τις μεταρρυθμίσεις στο προσκήνιο των θεμάτων της Ένωσης σε σχέση με τη Σερβία θα είναι πολύ σύντομα αργά. Ε, το να διατηρηθούν τα κεφάλαια 23 και 24 ανοιπτά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν είναι αποτελεσματικό Στη Σερβία χρησιμοποιούμε την έκφραση ότι όσο περισσότερα κεφάλαια ανοίγει η Σερβία, τόσο πιο λιγότερο δημοκρατική γίνεται. Μπορώ να σα το εξηγήσω. Στην Αλβανία, η Αλβανία μπορεί να κάνει κάποιε από τι βασικέ μεταρρυθμίσει, όχι πλήρω, αλλά υπάρχει, γιατί υπάρχει αντίδραση στι αλλαγέ από το κατεστημένο. Υπάρχει ισχυρή αντίδραση ε, μερικέ φορέ και ε, από μέσα από την κυβέρνηση και κυρίω σε σχέση και με το ε, οργανωμένο έγκλημα. Μπορώ να πω περισσότερα από αυτού η κυβέρνηση δεν ε, ε, αν δεν υποστηριχθεί θα ανατρέψει την πορεία. Το, το Κόσοβο έχει κολλήσει. Η υπάρχουσα ελίτ ε, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση δεν είναι διατεθειμένη να μετατρέψει ε, τον τρόπο διακυβέρνησης. Είναι ζωτική σημασία για το Κωσυφοπαίδιο να ολοκληρωθεί η ειρήνη με τη Σερβία και να περάσει ένα νέο κεφάλαιο για την οικοδόμηση του κράτους. Στην περίπτωση μη συμφωνίας οι υπάρχουσες ελίτ θα συνεχίσουν να για πολύ περισσότερο οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας, αν υπάρξει πλήρης λύση με τη Σερβία, θα επιφέρει αλλαγές στο Κόσοβο. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα είναι ευκολότερο να, πολυθεί, να περάσει μία, ένα συμβιβασμός από το να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή. Ε, το, το Κόσοβο έκανε πολλά στο θέμα του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά μόλις μόλις ε, ε, δεν μπορέσει να το πάρει, ε, όμω δεν μπόρεσε να το πάρει, υπήρξε κάποια πιστοχώρηση. Επίση, ε, ε, όσον αφορά του πολίτε, την κοινή γνώμη, βλέπουν ελάχιστε βελτιώσει από αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Το Μαυροβούνιο έχει επηρεαστεί θετικά στη Σερβία. Οι πολίτε ζουν χειρότερα όσον αφορά την ελευθερία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτο δικαίου. Η διαφορά ανάμεσα στο τώρα και στο ε, και στο παρελθόν είναι ότι δεν υπάρχουν πόλεμοι. Η ηγεσία έχει αποτύχει να ε, αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει κάποια ελπίδα. Μετά από πάνω από δεκαετία ε, απώλειας, μοιάζει απίθανη η επιστροφή καθεστώτος τύπου Γκρουεύσκη και η κυβέρνηση πλέον έχει δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στο Κόσοβο οι πολίτες όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για την επίλυση των θεμάτων με τη Σερβία. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πραγματικές και επηρεάζονται από το λόγο και τις συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει ευρύτατη ε, έλλειψη ικανοποίηση με την τρόπο διακυβέρνησης και επίσης πολλοί άνθρωποι ε, απομακρύνονται συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας και της Σερβίας. Ε, οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν χαμηλού επίπεδου, η παιδεία χαμηλού επίπεδου, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Ένα φίλο ε, που ε, πήρε διαζύγιο το 2008 και μόνο το 2018 κατάφερε να λυθεί η κατάσταση. Ε, επίσης, στη Βόρεια Μακεδονία πολλοί αισθάνονται ότι χάνεται έλεγχος. Σε κάποια στιγμή σε 5-10 χρόνια οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έχουν επιτύχει, ελάχιστοι θα έχουν μείνει στην περιοχή για να τις επιδιώκουν. Επίσης, ο λαϊκισμός. Στην Ευρώπη ο λαϊκισμός σημαίνει ότι στρεφόμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των μεταναστών. Στα Δυτικά Βαλκάνια σημαίνει ότι γινόμαστε εθνικιστές και ε, προωθούμε τις εθνικιστικές πολιτικές και τον συγκρουσιακό λόγο. Ε, αυτό έκανε ο Γκρουεύσκι στον περίοδο 2008-2016. Πιθανότατα θα το κάνει το Κόσοβο με τη Σερβία αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βλέπουμε ενδείξεις εντάσεων και μια ε, επιθυμία των ηγετών και των δύο κρατών να παραμείνουν στην εξουσία με κάθε τρόπο. Οι ελίτ των Δυτικών, Δυτικών Βαλκανίων έχουν κάνει καλού φίλους μέσα στην Ένωση. Τα κράτη-μέλη που είναι κατά τη διεύρυνση μιλάνε πολύ για το κράτο δικαίου. Αυτοί που υπονομεύουν το κράτος δικαίου στηρίζουν την διεύρυνση. Κάποιοι ηγέτε των Δυτικών Βαλκανίων κοιτάνε το μετέπειτα, την Ουγγαρία κλπ. Επίση. Ε, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις και η ελίτ έχουν χρήματα και πληρώνουν καλά τις δημόσιες υπηρεσίες, αυξάνουν τους μισθούς και έχουν δημιουργήσει πολλούς οπαδούς εντός του συστήματος, καθηγητές, δημόσιους λειτουργούς, ε, δασκάλους. Οι, οι υπάλληλοι είναι πιστοί και φοβούνται την αλλαγή, φοβούνται να χάσουν τις θέσεις τους και τους μισθούς τους. Αυτό αφήνει τη μεσαία τάξη σε δύσκολη κατάσταση. Τα χρήματα που παίρνει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει και να προωθήσει τις ε, μεταρρυθμίσεις είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν στα χέρια τους. Ε, ε, ε, το Κωσυφοπαίδιο και η Βόρεια Μακεδονία παίρνουν χρήματα τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που έχουν ήδη στα χέρια τους κυβερνήσεις. Κατά την άποψή τους τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι, αργούν να έρθουν, είναι άκαμπτα στους κανόνες τους και καθυστερούν το, η, απόδοσή τους. Ενώ ε, με την πολιτική οικονομία που υπάρχει η ελίτ ε, συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα κύματα και το σύστημα, χρήματα και το σύστημα λειτουργεί καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει τις δομές των ταμείων και τα προγράμματα που επικεντρώνονται στην υποστήριξη των αλλαγών εκ των κάτω για να επιτευχθεί η κοινωνική μετατροπή, η κοινωνική αλλαγή στα Δυτικά Βαλκάνια ε, καθώς υπάρχει αξιόπιστη προοπτική διεύρυνση της Ένωσης η προσέγγιση θα αλλάξει και αυτή. Τα ευρωπαϊκά ταμεία θα φτάσουν στην κοινωνία. Πρέπει να στηρίξουμε τη ζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις. Η Ιούλεξ του Κωσόβου θα πρέπει να φύγει, να αποχωρήσει και να ανοίξει την πόρτα για, μια, για νέες σημαντικές πρωτοβουλίες που δεν θα, ανακεφαλ, δεν θα επαναλαμβάνουν και θα ανακυκλώνουν τις προηγούμενες ή ε, παρόμοιες πρωτοβουλίες. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή και σωστή αξιολόγηση οι αποστολές τύπου Prime για όλες τις χώρες. Όπως και στη Μακεδονία θα πρέπει να είναι απολύτως δημόσιες συγκεκριμένες και να εμπλέκεται η κοινωνία. Ε, και να μετρώνται επίσης οι μεταρρυθμίσεις. Και τέλος, η, η πολιτική προσέλκυση της Ένωσης όταν υπάρχει λειτουργεί καλά. Η, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία προωθούν τις μεταρρυθμίσεις. Το Κόσοβο έχει εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά είμαστε ανάμεσα σε, ένα, σε μια χαλαρή έλξη και σε μια αυξανόμενη ε, δυσαρέσκεια των πολιτών ενώ οι ελίτ ε, δεν βλέπουν ε, δυσαρέσκεια προς τις ελίτ που δεν βλέπουν ακόμα τα πραγματικά ωφέλη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Μπορεί καλή μήπως να καταλήξει ότι οι κοινωνίες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν πολύ να προχωρήσουν για να μπορέσουν να ενισχύσουν τις ε, δημοκρατικές αυτές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Τώρα να δώσουμε το λόγο για ερωτήσεις προς τους ομιλητές μας. Ξεκινούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Παντζέρη. Δεν θέλετε το λόγο, εντάξει. Η κυρία Ίνετβελ, δεν έχει ζητήσει κάποιο το λόγο, απλώς ε, προσπαθώ να ξεκινήσω λίγο τη συζήτηση. Σόφι, παρακαλώ. Ναι, μία σύντομη ερώτηση, αφού άκουσα την τελευταία παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούμε εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα όχι μόνο στις χώρες προσχώρησης, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι η απάτη και η διαφθορά ε, που γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με το ζόρι την αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και δεν μπορεί να επαληθεύσει πώς ε, χρησιμοποιούνται τα χρήματα και από πού ξεκινάνε. Ποτέ όμως δεν άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι «Α, θα αλλάξουμε την προσέγγιση μας». Φαίνεται ότι συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο «business as usual» και νομίζω ότι αυτό που μόλις είπατε και το έχω ακούσει και στο παρελθόν κανονικά θα έπρεπε να οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Σόφη. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπουκίτσιο. ο οποίος μίλησε εκ μέρους Επιτροπής της Βενετίας. Έχω κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Αναφερόμαστε σε διεύρυνση και προσχώρηση και σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμάτων. Πρέπει από τη μια να αξιολογούμε τη σταθερότητα των λόγω χωρών και αφετέρου να θυμόμαστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με όλους. Ε, μιλάμε για τα Βαλκάνια και είναι καλή ευκαιρία εδώ να πούμε ότι ελπίζουμε ότι η διαμάχη ε, μεταξύ Μακεδονίας ή Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδος επιλύθηκε επιτέλους. Ε, αυτό το γεγονός μας υπενθυμίζει ότι τα λόγια, οι λέξεις και ο πολιτισμός έχουν σημασία και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ε, μια χούφτα κυβερνήσεων να το θέσει εν κινδύνο. Αναφέρεστε στον κίνδυνο μιας κατάστασης όπου μια πλειοψηφία κερδίζει τις εκλογές και εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που έχει να κάνει ό,τι επιθυμεί, ε, ανεξάρτητα από το κράτος δικαίου. Σε πολλές περιπτώσεις όμως ε, αναφέρεται κανείς στο δημόσιο συμφέρον και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό ακριβώ σας ρωτώ ως ε, νομικό. Πέρσι, για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, ε, υποβάλαμε ένα αίτημα κατά της Ουγγαρίας για να ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 7. Η Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σαφέστατα ότι αν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υποβάλει τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία 2 τρίτων. Ε, και εδώ το έχω και μαζί μου μάλιστα, έχω τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας. Και εκεί είναι σαφή τα πράγματα. Υπήρχαν τρεις δυνατότητες, υπέρ, κατά, αποχή. Πράσινο, κόκκινο και ε, κίτρινο. Και δεν γνωρίζω να υπάρχει πουθενά κανένα άλλο πολιτικό οργανισμό παγκοσμίω, είτε σε χώρα, είτε σε οργανισμό, είτε σε ε, διεθνέ κοινοβούλιο, να υπάρχει δυνατότητα ε, σταθμισμένη πλειοψηφία που οδήγησε σε αυτό το οποίο διαπιστώσαμε εδώ σήμερα. Υπάρχουν μια σειρά Ήθελα να μιλήσω με μια σειρά από περιογνωμόνε με το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Όχι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είπανε κάποιοι ότι δεν θα ληφθούν οι ψήφοι τη αποχή σε αυτή την περίπτωση κατά τη Ουγγαρία. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό, γιατί έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι αποχέ. Γνωρίζετε λοιπόν εσείς κανένα παράδειγμα στο οποίο η ειδική πλειοψηφία οδήγησε σε να, να μην ληφθούν υπόψη οι αποχές. Υπολογίστηκε δηλαδή η ειδική πλειοψηφία χωρίς αποχές. Τώρα, η κύρωση της συνδίκης της Κωνσταντινούπολης και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το βλέπουμε αυτό και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία, διαθέτουν συνταγματικό δικαστήριο το οποίο απεφάνθη ότι η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης δεν συνάδει με το οικογενειακό δίκαιο του συντάγματος της χώρας στη Βουλγαρία. Βλέπουμε λοιπόν συνεχώς να πιέζεται η χώρα αυτή ώστε το Κοινοβούλιο ε, και η κυβέρνηση να ε, προωθήσουν ε, και να αναρέσουν την απάντηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας και δεν θα πρέπει να επιτρέπει στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια να κάνουν ό,τι επιθυμούν όταν υπερβαίνουν το Σύνταγμα. Και τελικά βλέπουμε τι γίνεται. υπάρχουν μια σειρά από στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα. Εσείς είπατε ότι υπάρχουν χώρες οποίε υπάρχει μια πλειοψηφία που δεν μπορεί να επιβάλλει τα πράγματα στη μειοψηφία, δεν βλέπετε να γίνεται ακριβώ το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει η ίδια έλλειψη ασφάλεια δικαίου, διότι... Ε, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Τα ίδια δεν συμβαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Πέτριλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 15 χρόνια έγινε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Θεσσαλονίκη που έδωσε μια ευρωπαϊκή προοπτική στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ακόμα όμως η κατάσταση είναι στο ναι μεν αλλά. Με την ε, συνήθη διάγνωση. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να έχουμε μία ένωση με δύο διαφορετικές ερμηνείε του κράτους δικαίου. Οπότε η ερώτησή μου στα μέλη του πάνελ είναι αν έχουν κάποια ιδέα για το πώς μπορεί να κινηθεί η διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριε Νταμόφ. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Ωραία. Ναι. Κάτι. Οπωσδήποτε. Ε, είπε η κυρία Ινετφέλτ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, βεβαίω. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που έθεσε η κυρία Ινετφέλτ και βεβαίω υπάρχει ανάγκη να ε, προσαρμόζουμε συνεχώς τα μέσα μας για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε. Και το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε σχετίζεται με τον στόχο μας που είναι να στηρίξουμε τις ε, χώρες οι οποίες είναι σε μια διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικότερος πολιτικός στόχος είναι σαφής. Είναι ότι οι χώρες αυτές, όπως αναφέρει και η απόφαση της ε, Θεσσαλονίκης, να γίνουν ε, στο μέλλον κράτη-μέλη. Έχει γίνει τίποτα έκτοτε. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή συνεχής ε, και όσον αφορά τα μέσα με τα οποία εργαζόμαστε και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Τα ανέφερα λίγο στην εισαγωγή μου. Οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Θα πω μόνο ότι νομίζω τώρα έχουμε εκθέσει επαρκώς την προσέγγισή μας ε, για την στρατηγική στα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε από την πολιτική πλευρά είναι ξεκάθαρα σαφές ότι η επιλογή αυτή αφορά τις ε, εν λόγω χώρες αν θέλουν να προχωρήσουν ή όχι. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τις ε, στηρίξουμε και έτσι όπως το έχουμε ε, παρουσιάσει στην στρατηγική είναι υπομορφή 35 συγκεκριμένων 53 συγχωρείτε, συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν και το κράτος δικαίου. Οπότε το ένα είναι αυτό, ένας νέος τρόπος άλλο είναι το πώς εργαζόμαστε στις διαπραγματεύσεις. Και εδώ πέρα νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αλλάζουμε κάθε χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Οπότε, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από τα βασικά και υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία προόδου στα κεφάλαια 22-23 και στις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις. Αυτό κάνουμε. Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο που ανέφερε ένας ε, συνάδελφος εδώ το πώς μπορούμε να εργαστούμε περισσότερο στις χώρες αυτές για να ξεκαθαρίσουμε το τι κάνουμε και το τι προσδοκίες έχουμε. Και εδώ πέρα συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα όταν μιλάμε για την δημόσια διπλωματία, να ενεργοποιηθούμε, να είμαστε σαφείς επί τόπου για το ποιες είναι οι συνέπειες της αδράνειας, αλλά και στο τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνουν αυτές οι χώρες. Και είναι ξεκάθαρο αυτό όσον αφορά την κατεύθυνση της υπαναχώρησης. Ε, και βέβαια, αν δείτε τις δηλώσεις Κομισιόν, θα δείτε ότι είμαστε πολύ ενεργοί στο ε, πεδίο αυτό, όταν δεν υπάρχουν κάποιες ε, δράσεις και κάποιες εξελίξεις, κάτι το οποίο δυστυχώς συνέβη τις τελευταίες δύο μήνες. Νομίζω ότι έτσι απάντησα και για τον, την δυναμική της διαδικασίας. Τέλος να πω ότι Βεβαίως, εγώ θα έλεγα από την πλευρά της ε, Κομισιόν ε, και του Κοινοβουλίου θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε το ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποια στήριξη δίνουμε στις ε, χώρες. Σε τελική ανάλυση αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από τις πολιτικές ελίτ, την κοινωνία των πολιτών, τους ρόντες στις χώρες αυτές ε, μια απόφαση που θα λάβουν αυτοί και μετά θα κάνουν και τα απαραίτητα βήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, σύντομες αντιδράσεις στα σχόλια και τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Πρώτα από τον κύριο Μποκίκιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Γιούρεκ, αν δεν κάνω λάθος. Συμφωνώ μαζί σας. Υπογραμμίσατε τη σημασία του παράγοντα σταθερότητα στη διαδικασία ένταξης. Φυσικά είναι σημαντική η σταθερότητα. και το ευτυχές τέλος της σύγκρουσης ε, Βόρειας Μακεδονίας Ελλάδας είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Θα ήθελα στο άμεσο μέλλον να δω και άλλες τέτοιες συγκρούσεις να επιλύονται για να ε, διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης. Όσον αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, από το σεβασμό του κράτους δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικό μου θέμα να τοποθετηθώ επ, αυτού. Συμφωνώ ε, για τη σημασία της συμφωνίας ε, των συμφωνιών της Βουλγαρίας που αναφέρατε και αυτό που έκανε, αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρετε ποια είναι η θέση μου. Η, αποφάση των κοινωνικών συμφώνων, το... η συμφωνία, η... ουσιαστικά οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων πρέπει να γίνονται σεβαστές και όταν ε, οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα έχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ κύριε Μπουκίκιο. Και δύο σύντομες απαντήσεις από τον κύριο Κμέτριτς. Αν θέλετε φυσικά. Ναι, μπορώ βεβαίως. Αν δεν θέλετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω όσον αφορά τη σταθερότητα. Ή μάλλον πρώτα-πρώτα για τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς γίνονται δεκτά στην περιοχή. Διότι προφανώς αυξάνεται η σύγχυση από για το τι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Διότι αν ζεις εκεί, τα, τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν για παράδειγμα έχουμε ένα Πρωθυπουργό ο οποίος κατηγορείται για την παραβίαση ε, του κράτους δικαίου ε, στην Βόρεια Μακεδονία και μετά λαμβάνει άσυλο ε, στην Ουγγαρία, είναι λίγο συγκεχημένα. Και εδώ φυσικά είναι σαφές τι γίνεται με τα μηνύματα και εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στα θέματά σας. Θα πρέπει να έρχονται με πιο σαφή τρόπο, να είναι πιο ξεκάθαρα και να περιλαμβάνουν και τα διάφορα θέματα, γιατί δάλλως κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτούς που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τους θειασότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ακριβώς της έλλειψης αντίδρασης για την παρούσα υποχώρηση της δημοκρατίας στην περιοχή. Αν χάσουμε λοιπόν αυτές τις δημοκρατικές φωνές, Ποιο θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Απλώς ε, κοιτούσα λίγο το πρόγραμμα να δω ποιος θα απαντήσει ε, στη, στις απαντήσεις που λάβαμε. Δεν ήθελα ε, να προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι λίγα τα μέλη εδώ. Θέλει κάποιο να δώσει μια σύντομη απάντηση. Κύριε Σίτη, μήπω θέλετε εσείς, αλλά σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, αυτό το καλοκαίρι Υπήρχε συζήτηση για τη διαδικασία απελευθέρωσης ε, των ε, υποχρεώσεων θεωρήσεων διαβατηρίων. Ε, η απάντηση ήταν δεν εμπιστευόμαστε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια μπορεί να εμπιστευτεί. Και σε αυτή τη σύγχυση αναφερόταν ο συνάδελφος. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία θα πρέπει να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό ουσιαστικό για την περιοχή. Δεύτερον, επενδύσεις ε, για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας το συντομότερο δυνατόν. Το πολιτικό βάρος ε, των κρατών μελών είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσουν τα πράγματα. να υπάρχουν ε, ε, ε, βανάγνωστες εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγχειρίδια για κάθε χώρα και να μεγαλώσει η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, να καλέσετε κάθε μεγάλη ομάδα για να συνεργαστούν μαζί σας. Και επίσης η επιχειρηματικό κοινότητα είναι διατεθειμένη παρά τα όσα συμβαίνουν με την πολιτική κατάσταση και το κράτος δικαίου, επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στο Κωσυφοπέδιο, στην Αλβανία, στην ε, Βόρεια Μακεδονία και στη Σερβία. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλος ο αριθμός ε, των ε, συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρατηρήσεις. Πριν ζητήσω από τον κύριο Κούκαν να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, εξ του κυρίου Κουσόη και του υποφαινομένου, να ευχαριστήσω τα μέλη ε, των επιτροπών που ήρθαν εδώ. Θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερους. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι λόγοι, είμαστε στο τέλος της θητείας, είναι Δευτέρα, έχουμε πολλούς λόγους, αλλά φυσικά σε καμία περίπτωση αυτό δεν υπομονωμεύει το, τη σημασία του θέματος που συζητούμε. Βλέπω εδώ ένα μακρύ κατάλογο εισηγητών εκ μέρους της Επιτροπής μας για τα θέματα κράτους δικαίου. Η Σόφι Ινετβέλντ ε, προεδρεύει στην ομάδα για το κράτο δικαίου και έχουμε και πάρα πολλού συγητέ ε, για τι εκθέσει αναχώρα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, έχει γίνει πολλή δουλειά για τα θέματα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και πολύ έντονε οι επαφέ μεταξύ των επιτροπών μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν αντανακλάται σήμερα όμω στον αριθμό των μελών που είναι παρόντα εδώ. Να ευχαριστήσω όμω του ομιλητέ που ε, προσέδωσαν στο θέμα τη σημασία που του αξίζει. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κουσό που ήταν εδώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κούκαν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας ε, της ε, ΑΦΕΤ, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Δυτικά Βαλκάνια. Θα συνοψίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι τηλεγραφικός στα συμπεράσματά μου. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι εκτιμώ τους εμπειρογνώμονες και ιδίως το γεγονός ότι στις παρεμβάσεις τους αναφέρθηκαν βάση πραγματικής ε, πολιτικής ζωής και πραγματικής πολιτικής κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην κάθε χώρα. Δεν ήθελαν ε, να μας εντυπωσιάσουν ε, με εξεζητημένες αναλυτικές θεωρητικές αναλύσεις, αλλά μίλησαν βάσει όσο όσων συμβαίνουν επί τόπου και αξιολόγησαν την κατάσταση ως έχει. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους συναδέλφους που ήρθαν στη συζήτηση και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι είχαμε την ευκαιρία να γίνει αυτή η ενημέρωση πριν ολοκληρωθεί η παρούσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το προσυζήτηση θέμα βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι έλαβαν το λόγο συμφωνούν ότι το κράτος δικαίου είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στη διαδικασία ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τόνισαν φυσικά όλοι ότι αυτό αποτελεί τη βάση για να γίνει κάποιος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε σημασία στο κράτος δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε τη σημασία του και να συνεχίσουμε να το τονίζουμε στους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παραμείνουν ε, με αποφασιστικό τρόπο στα αιτήματά τους για το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των πολιτών και το, την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών στην περιοχή. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω αυτό που είπε και ο κύριος ε, Μπουκίχο εδώ, τα θέματα του κράτους δικαίου πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν το σθένος ε, και τις δυνατότητες να εξηγήσουν στους πολίτες τους ότι τα θέματα αυτά δεν ε, τα συζητούμε απλώς για χάρη των Βρυξελών. Οι κυβερνήσεις δεν κάνουν πράγματα για να ικανοποιήσουν τις Βρυξέλλες, αλλά για μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες της χώρας. Μπορεί να είναι δύσκολο μεν αυτό, αλλά πρέπει να γίνει για να πιστούν οι πολίτες ε, και να κατανοήσουν τι ακριβώς ε, εννοούμε. Θα πρέπει να γίνει μια ρεαλιστική αξιολόγηση για το πού βρισκόμαστε στη διαδικασία της διεύρυνσης. Είναι σαφές ότι χωρίς ε, μια απτή διαδικασία στο κράτος δικαίου που περιλαμβάνονται και στα κεφάλαια 23 και 24, περαιτέρω διαδικασία ένταξης ε, δεν θα μπορέσει να υπάρξει. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ε, άκουσα κάποιες επικρίσεις από τους δύο συναδέλφους ε, και κάποιες διαμαρτυρίες αν θέλετε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί και πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατανοητά όλα αυτά και εγώ πάντα λέω ότι η διαδικασία διεύρυνσης είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των εταίρων μας και ημών. Και αν το ζητήσουμε να μας δώσουν αποτελέσματα και φέρουν τα αποτελέσματα, τότε είναι καθήκον μας να κάνουμε και εμείς το αντίστροφο. Εάν ε, μας δώσουν αποτελέσματα και εμείς προβάλλουμε νέες απαιτήσει, τότε χάνεται η αξιοπιστία μας. Πρέπει λοιπόν να το δούμε έτσι το ζήτημα. Και επίσης συμφωνώ με τον κύριο Ντάνιτς, ο οποίος είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ ε, αυστηροί και να λέμε στους εταίρους μας ότι πρέπει να τηρούνται πλήρως τα κριτήρια και οι απαιτήσεις. Ιδάλλως δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις ή πιο σύντομες οδοί. Αν εξετάσει κανείς την περιοχή, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν θα επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες και να μιλήσω για κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά σε γενικές γραμμές, και το ακούσαμε αυτό και ε, από τους ομιλητές, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημάδια επαναχώρησης, ιδιαίτερα σε κάποιες πτυχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι αλήθεια ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος ήταν ε, υψηλή προτεραιότητα σε κάθε χώρα της περιοχής, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλουν. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί ε, το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες συστάσεις για το κράτος δικαίου, ε, κυρίως για μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένες χώρες. Τα κεφάλαια 23 και 24 είναι ο πυρήνα τη διαδικασία ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, διότι αφορούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Πρέπει λοιπόν να τους υπενθυμίσουμε ότι είναι ακόμα πολύ επίκαιρα. Τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν ποιος και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα εδώ, επί τη ευκαιρία, να αναφέρω το πρώτο από τα κριτήρια, διότι είναι πάντα καλό να το υπενθυμίζουμε. Αναφέρεται στη σταθερότητα των θεσμικών οργάνων που εγγυούνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Χωρίς σαφέ μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ότι το μήνυμα θα αποτελέσει το κληροδότημα της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το δεύτερο ήμιση του 2019 θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστούμε τους ομιλητές και αυτούς οι οποίοι οργάνωσαν την ακρόαση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους.